σύμφωνα με το άρθρο 149 του κανονισμού το τελικό σχέδιο της, ε, των εργασιών έχει διανεμηθεί. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις. Για την Τρίτη, θα ήθελα καταρχήν να σας αναφέρω το εξής. Δεδομένη τη σημερινή κατάσταση όσο έχει διαμορφωθεί και σε επαφή με τα άλλα θεσμικά όργανα προτείνω τις εξής αλλαγές στην ημερήσια διάταξη ο κύριος Τούσκ για αύριο το μεσημέρι θα έχει μια έκτακτη σύνοδο που συνεκάλεσε της Ευρωζώνης. Γι' αυτό το πρώτο σημείο την Τρίτη το απόγευμα θα είναι η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η προπαρασκευή του προγράμματος εργασιών για το 2016. Και αυτό αντί της μέχρι τώρα στην ημερήσια διάταξη των ε, τελικών ε, συμπερασμάτων ε, του Συμβουλίου για την Σύνοδο του Ελληνής Κατάστασης στην Ελλάδα. Ανταυτού σας προτείνω την Τετάρτη το πρωί ως δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη να είναι η δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της, του Ιουνίου και για την σημερινή επίκαιρη κατάσταση στην Ελλάδα. Και αυτό να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη. Αυτό το σημείο αντικαθιστά την δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προπαρασκευή του προγράμματος εργασίας. Και αν εγκρίνεται αυτό, τότε για την Τρίτη έχει επισπευστεί αυτό το θέμα. Και εκτός τούτου μου ζητήθηκε λόγω του ότι υπάρχουν πολλές παρεμβάσεις την ώρα της ψηφοφορίας να ξεκινήσουμε στις 13 ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο για τις παρεμβάσεις για τη συζήτηση. Κάτι θέλετε να πείτε για την Τετάρτη κύριε Φεχόστατ. Παρακαλώ. Ναι, είναι η μόνη δυνατότητα η συζήτηση που προβλέψαμε για την Ελλάδα να αναβληθεί για την Τετάρτη μετά την διάσκεψη. Όμως πρέπει να σας πω ότι ο πρόεδρο τη Επιτροπή και ο πρόεδρο του Συμβουλίου θα είναι αλλά πρέπει και ο κύριο Τσίπρας να είναι για να έχουμε μια πλήρη συζήτηση και ο κύριο Ντάισεμπλουμ από το Eurogroup να είναι επίση παρόν. Γιατί είναι τρελό να συζητήσουμε για την κατάσταση στην Ελλάδα χωρί τον Πρωθυπουργό τη Ελλάδα εδώ παρόντα σε αυτό εδώ το μικύκλιο. Είναι, πρέπει να σας πω, ένας από τους πολιτικούς μου αντιπάλους είναι ο κύριος Ορμπάν, αλλά όταν μιλάμε για την Ουγγαρία είναι παρόν ακόμα και αν διαφωνώ μαζί του, είναι παρόν. Οπότε νομίζω ότι αν θέλουμε πραγματικά να συζητήσουμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο, αν θέλουμε πραγματικά να συζητήσουμε για πιθανέ ε, λύσει, τότε και ο Έλληνα Πρωθυπουργό πρέπει να είναι παρόν μαζί με τον κύριο Ντάισεμπλουμ που είναι ο πρόεδρο του Eurogroup. Σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φερχόστατ, συμμερίζομαι το αίτημα σε σχέση με αυτό. Για την τρίτη τώρα και Τετάρτη το πρωί. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να παρέμβουν. Παρακαλώ εσείς κυρία. Η κυρία Χάμς για την ανακοίνωση αυτή θέλετε να κάνετε. Είναι ένα αίτημα του κυρίου Φερχόφστατ που οπωσδήποτε ήθελε να υποστηρίξει το Κοινοβούλιο Κατά τις τελευταίες εβδομάδες επανειλημμένα προσπαθήσαμε πριν από τις συνόδους κορυφής και πριν από τις αποφασιστικές ε, διασκέψεις να συζητήσουμε από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να καταλήξουμε σε αποφάσεις. Πάντα ζητούσαμε και με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης να γίνουν διαπραγματεύσεις. Απορρίφθηκε το αίτημά μας. Ανταυτού εσείς τοποθετηθήκατε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήρθε επιτέλους η χρονική στιγμή να διεξαχθούν άμεσα αυτές οι συζητήσεις. Πρόεδρος, κυρία Χάμς, δεν έχω γνώση περί τίνος κάνετε λόγο τώρα εσείς. Δεν το γνωρίζω. Αν είσαστε παρακαλώ τόσο ευγενείς να μου το... Αν δεν ακούτε ούτε καν τις απαντήσεις μου, τότε εντάξει, κύριε Φαντάρ. Κυρία Χάμς, ήθελα να σας δώσω μια απάντηση, αλλά τώρα πια πέρασε η ώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Από διάφορες πλευρές ακούσαμε για το δικό σας ρόλο στην εκστρατεία υπέρ του ναι στην Ελλάδα. Και λέμε τώρα για τη συζήτηση που θα γίνει την Τετάρτη εδώ. Οπότε, ακούσαμε την πρόταση να ακουστούν και άλλοι. Και εσείς είχατε κάποιο ρόλο στην εκστρατεία του ναι, οπότε θα ήταν υπεύθυνο τώρα να τοποθετηθείτε για την Ουγγαρία ήτανε αλλιώς τα πράγματα όταν πρόκειται για την Ουγγαρία τότε πολύ συχνά εμείς εκφραζόμαστε με μια πλειοψηφία. Εδώ όμω δεν είχαμε τη δυνατότητα να εκφραστούμε. Το κάνατε εσείς υπέρ του ναι χωρίς εμείς να έχουμε τη δυνατότητα να εκφραστούμε. Προτείνω λοιπόν στη συζήτηση αυτή της Τετάρτης και εσείς να έχετε τη δυνατότητα να εκφραστείτε για το ναι και άλλοι για ό,τι πιστεύουν στη συζήτηση της Τετάρτης. Ευχαριστώ. Ε, δεν έχω άλλη δυνατότητα από τον κύριο Ντάισερμπλουμ και τον κύριο Τσίπρα να γνωστοποιήσω απλώς το αίτημα του Ευρωκοινοβουλίου. Εντάξει, θα το κάνω. Αυτό ζητήθηκε να κάνω. Δεν έχω την εντύπωση ότι όλοι τοποθετήθηκαν επ' αυτής της επιθυμίας. Αλλά θα το εκθέσω. Αυτό εντάξει. Ερωτώ τώρα για την τρίτη. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να παρέμβουν. Για την ημερήσια διάταξη της Τρίτης. Για την Τρίτη, ο κύριος Γλέζος είχε ζητήσει να παρέμβει σε ένα αίτημα που είχε για την ημερήσια διάταξη που αυτό, εκείνος και άλλοι 51 ευρωβουλευτές ήθελαν να καταθέσουν για μια δήλωση της Επιτροπής και του Συμβουλίου για τις γερμανικές επανορθώσεις. Έχετε τον λόγο κύριε Γλέζο, παρακαλώ. Ναι, αυτό ακριβώς ήθελα να καταθέσω αγαπητέ Πρόεδρε. Εάν πρόκειται να γίνει η συζήτηση σήμερα σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, αν πρόκειται να δεχτεί το Κοινοβούλιο να συζητήσουμε το θέμα των οφειλών της Γερμανίας βάσει του κανονισμού καταθέσαμε 50 ευρωβουλευτές, 51 ευρωβουλευτές την αίτηση. Και ήθελα να ρωτήσω την άποψή σας πώς θα διεξαχθεί η διαδικασία για το θέμα. Ένα αυτό. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους ευρωβουλευτές να μην τους κακοφανεί θα υπερασπιστώ τον α, πρόεδρό μας τον ε, Μάρτιν Σούλτς περίεργο ε, θα τον υπερασπιστώ όμως διότι η αγάπη του για την Ελλάδα εκφράστηκε επανειλημμένα αλλά ο ελληνικός λαός απέρριψε την πρότασή του να είναι μονάρχης διοικητής των δανειστών στην Ελλάδα. Επειδή όμως το αίτημά του το γνωρίζω για την αγάπη του για την Ελλάδα, θα του πρότεινα να έρθει στην Ελλάδα, να γίνει πολίτης της Ελλάδας και να ε, μπει σε οποιοδήποτε από τα κόμματα θέλει και εγώ θα τον υπερασπιστώ και θα τον υποστηρίξω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γλέζο. Το αίτημά σας εμπρόθεσμα κατατέθηκε και άλλοι 51 ευρωβουλευτές προσυπέγραψαν. Ο τίτλος είναι «Δήλωση της Επιτροπής» καθότι με ενημέρωσαν και του Συμβουλίου και τη Επιτροπή, αλλά όχι, μόνο της Επιτροπής, Δήλωση της Επιτροπής για τι ε, ε, για τις γερμανικέ οφειλέ. Κάποιο ε, για το αίτημα αυτό, κυρία Τσίμερ, εσείς παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, θέλω να σα παρακαλέσω να γίνει δεκτό το αίτημα του κυρίου Γλέζου. Έχουμε εδώ ένα ζήτημα ενώπιόν μας που αφορά πάμπολους ανθρώπους στην Ελλάδα, εδώ και δεκαετίες τους απασχολεί και που με τις συμβάσεις και συνθήκες του 1991 δεν έχει διευθετηθεί και είναι κατεπηγόντως αναγκαίο, θεωρούμε, έναντι του ευρωπαϊκού λαού να δειχθεί ο σεβασμός ε, με μια συζήτηση που θα διεξαχθεί εδώ. Μπορεί κανείς να πει ότι αυτό ίσως είναι ένα διμερές θέμα μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Αλλά αυτά τα θέματα αφορούν και το κλίμα και την ατμόσφαιρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το λέω αυτό συνειδητά ως Γερμανίδα Ευρωβουλευτήνα. Ότι θεωρώ δηλαδή και πιστεύω ότι εδώ υπάρχει μια ευκαιρία να έχουμε έναν ισοδίκαιο, τίμιο τρόπο να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα που εκκρεμούν εδώ. Και δεν πρόκειται για χρηματικές εξοφλήσεις, αλλά για την αναγνώριση ότι πραγματικά πρόκειται για θέματα που δεν έχουν επιληθεί και πρέπει να έρθουμε σε επαφή και να συζητήσουμε ανάμεταξύ μεταξύ μας για αυτό το ζήτημα. Πρόεδρος, θέλει κάποιος να λάβει τον λόγο κατά του αιτήματο αυτού. Κύριε Πρέντα, παρακαλώ. Oui, monsieur le président. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό το τσίρκο που εξάγουν οι κομμουνιστές της Ελλάδας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε πίσω, να σταματήσουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για να κάνουμε ό,τι να είναι με αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό είμαι κατά αυτή της πρότασης των κομμουνιστών που έχουν φέρει την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση Äh, ένας Ευρωβουλευτής τοποθετήθηκε υπέρ, ένας εναντίον του αιτήματο. Θα θέσουμε το αίτημα σε ψηφοφορία. Όσοι είναι υπέρ να σηκώσουν το χέρι παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε το αίτημα. Περνάμε τώρα στην Τετάρτη. Θέσατε το έτοιμά σας για την Τετάρτη ήδη. Άλλοι θέλουν να παρέμβουν για την Τετάρτη. Δεν θέλουν να παρέμβουν άλλοι. Περνάμε λοιπόν τώρα στην Πέμπτη. Ζήτησε η έκθεση για την τεχνολογία και να, να αναβληθεί για το Σεπτέμβριο. Για να επιχειρηματολογήσει έχει τον λόγο καταρχήν η κυρία Σάκε παρακαλώ. Α, κυρία συγγνώμη. Έχετε τον λόγο, um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και συναδελφοί. Μετά από συνεργασία σε πολύ καλό τμήμα κλίμα για τα θέματα τη τεχνολογία και πώ επηρεάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίω, φαίνεται ότι χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο να διευκρινίσουμε κάποιε ασάφειε και κάποιε διαφορέ μεταξύ των ε, ε, πολιτικών ομάδων και βάσει του άρθρου 152 παραγράφου 1 θα ήθελα να ζητήσω να αναβολή μέχρι το Σεπτέμβριο. Υπέρ του αιτήματο ο κύριο Βάιντεν, υπέρ παρακαλώ. Θέλω να προσθέσω και εγώ τη φωνή μου σε αυτό. Είχαμε επικοδομητικέ συζητήσεις ανεφίσαν πρόσθετα προβλήματα. Είναι ένα σημαντικό θέμα, πρέπει να έχουμε περισσότερο χρόνο γι' αυτό και εγώ θα ήμουν υπέρ του να αναβάλουμε μέχρι την επόμενη σύνοδό μα του Σεπτεμβρίου τη συζήτηση. Άλλοι που θέλουν να παρέμουν δεν υπάρχουν. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν να αναβληθεί για το Σεπτέμβριο, να σηκώσετε το χέρι σας. Κατά αποχές εγκρίθηκε και αναβάλλεται λοιπόν η έκθεση αυτή η ομάδα Άλντε ήδη μέσω του κυρίου Γιάκοβ είχε προαναγγείλει ότι είχε σκοπό να διεξαχθεί μια συζήτηση <clears throat> με ψήφισμα για την πέμπτη ως πρώτο σημείο στην ημερησία διάταξη. Κύριε Γιάκοβ και τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η επιθυμία της ομάδας ε, των φιλελευθέρων είναι η Σρεμπρένιτσα και η καταστροφή της Σρεμπρένιτσα να ε, τύχει ε, μιας κατάλληλη τιμή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Όπω κάνατε και εσεί με την ενεκτήρια ομιλία σα, κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό και εμεί θα θέλαμε ευρωβουλευτέ να είμαστε ενωμένοι σε αυτό το ψήφισμα ω φόρο τιμή στα θύματα τη Ρεμπρένιτσα και των υπολείπων θυμάτων των Βαλκανικών χωρών και γι' αυτό ακριβώ το λόγο θα θέλαμε να υπάρχει αυτό το ψήφισμα το συντομότερο δυνατόν και γι' αυτό ακριβώ θα ήθελα να σα ζητήσω κυρίε και κύριοι ευρωβουλευτέ, να υποστηρίξετε την πρόταση και να υπερψηφίσουμε αυτό το ψήφισμα την Πέμπτη το πρωί. Ευχαριστώ. Κύριος Πλέκενστάιν, παρακαλώ υπέρ του αιτήματο. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε υπέρ του αιτήματο. Ακόμα και αν στη διάσκεψη των Προέδρων για κάποιους καλούς θετικούς λόγους μια άλλη οδός επελέγει. Πιστεύουμε ότι τα δεινά τα οποία υπέστησαν χιλιάδες άνθρωποι πρέπει να αξίζουν ώστε να έχουμε μια νυφάλια σε βάθος συζήτηση όπως πρέπει και αυτό το αξίζουν τα άτομα που δολοφονήθηκαν εκεί και απεβίωσαν και αξίζουν να τύχουν αυτή τη συζήτηση. Πρόεδρος, κάποιος κατά του αιτήματο, κύριε Φανόρντεν παρακαλώ. Uh, thank you very much, uh, President. Ευχαριστώ. Είμαστε απόλυτα υπέρ της συζήτησης αυτής την Πέμπτη. Αύριο όμως οι Ευρωπαίοι συντηρητικοί αύριο το βράδυ έχουμε όλο το βράδυ εκδηλώσεις για να τιμήσουμε ακριβώς τα θύματα. Οπότε όποιο θέλει μπορεί να έρθει. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει κανείς όμως που να είναι κατά του αιτήματο, εντάξει. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε επί του αιτήματο. Όσοι είναι υπέρ, παρακαλώ να σηκώσετε το χέρι σας κατά άποχες νομίζω η πλειοψηφία ήταν εκείνη που ήταν υπέρ η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών κατάθεση για ψηφίσματα προθεσμία για την κατάθεση ψηφισμάτων είναι αύριο 10 η ώρα το πρωί Κοινέ προτάσει ψηφίσματο Τετάρτη 12 το μεσημέρι. Και για τροπολογίε σε αυτέ τι κοινέ προτάσει ψηφίσματος προθεσμία Τετάρτη 8 <clears throat> Ιουλίου 13.00. Και θα ψηφίσουμε την 5η ε, 9 Ιουλίου. Εντάξει, και έτσι λοιπόν εγκρίθηκε η μερίσια διάταξη της περίοδου συνόδου. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Για διαδικαστικό, εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε η ελληνική είναι εκείνο το οποίο την χάνει της ε, προσοχής μας και θέλω να στρέψω την προσοχή στο εξής. Κάποιος που ήρθε πριν από 80 χρόνια σε αυτόν τον κόσμο, κάποιος που τον γνωρίζετε και τον ε, εκτιμάτε για την ανεκτικότητά του και την προσπάθη, τις προσπάθειές του για την ειρήνη και είναι ο Δαλάι Λάμα, ο Παναγιώτατος Δαλάι Λάμα που γίνεται 80 ετών σήμερα και τις ε, δραστηριότητες που έχει αναλάβει και του εύχομαι όλα τα καλά για τα γενέθλιά του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, ε, ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή